Πάμε στο επόμενο θέμα, συνάδελφοι. Έχουμε αυτήν την μελέτη που αναθέσαμε για το Συμβούλιο που ονομάζεται από τη Συνέλευση Πρεσβευτών σε πραγματικό κοινοβουλευτικό σώμα και έχουμε κοντά μας τον καθηγητή Ολιβιέ Ρόζενμπεργκ. Um, uh, without further ado, I will just give you the floor. Να σας δώσω το λόγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Yes. So, can go? Yes, Thank you, Mrs. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οπότε να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση που μα ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, είναι το, το, το, το, το πώς μπορούμε να φέρουμε περισσότερο κοινοβουλευτισμό στο Συμβούλιο. Και έβαλα τον τίτλο αυτόν που είπατε «Το Συμβούλιο από Συνέλευση Πρεσβευτών σε Πραγματικό Σώμα Κοινοβουλευτικό». Και κάποιος φιλόσοφος Ιρλανδός είχε πει το 1974 ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι μια συνέλευση πρεσβευτών. Αλλά οι πρεσβευτέ ε, φροντίζουν κάποια συμφέροντα, ενώ, ενώ το κοινοβούλιο ασχολείται με άλλο πράγμα, ασχολείται με κάποιε απόψει. Ε, βέβαια και συμφέροντα, αλλά γίνονται συμβασμοί κλπ. Οπότε θεώρησα ότι πρόκειται για το Συμβούλιο, γιατί αυτό ακριβώ γίνεται σε επίπεδο κορεπέρ, σε ομάδε εργασία ακόμα και σε το επίπεδο του Συμβουλίου Κορυφής. Βεβαίω και εκεί προέρχονται τα συμφέροντα των κρατών μελών. Οπότε για να δούμε. Μπορεί, είναι δυνατόν να δώσουμε εκεί μια μορφή, ένα σχήμα κοινοβουλευτικό. Να δούμε πρώτα πρώτα ποια είναι η δομή του Συμβουλίου. Υπάρχει ένα τέτοιο σχήμα κοινοβουλευτικό ε, στο οποίο μπορεί να χωρέσει, να συντεριάξει το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να, κοινοβουλευτοποιηθεί και η απάντησή μου σύντομα είναι καταφατική ναι ναι είναι δυνατό υπάρχει δεδομένο τέτοιο σχήμα ε, είναι περίπλοκο ναι επίσης ε, και όχι γιατί υπάρχει συμπληρωματικότητα όσον αφορά το αν συντεριάζει το Συμβούλιο και επίσης ε, υπάρχει περιπλοκότηση γιατί απαιτείται μια διαφάνεια ε, στις εργασίες ενός ε, κοινοβουλίου να ποιο είναι το πρότυπο, το, το, το, το καλούπι του γενοβουλίου και Επίσης έχουμε τις ε, δραστηριότητες ενός κοινοβουλίου, την οργάνωσή του, επίσης τις διαδικασίες που γνωστές ή όχι, όσον αφορά τη συζήτηση, όσον αφορά τη διαφάνεια, αυτά και όχι μόνο αυτά και άλλα στην εκθεσή μου προσπάθησα να κάνω κάποια αξιολόγηση σε αυτά τα 13 στοιχεία για το Συμβούλιο και απαντώ καταφατικά ή λέω καταφατικά κάθετος, όχι κάθετος ναι. Και εδώ υπάρχουν τα τρία βασικά στοιχεία. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν ε, κοινοβουλευτική δομή, φύση. Ε, υπάρχει αντιφάσκη ουσία τους. Ας πούμε όσον αφορά τα μέλη, όλοι σαν κοινοβούλιο έχουν ε, ίσα δικαιώματα ψήφου. Αυτό δεν ισχύει ε, στο Συμβούλιο. Και βέβαια υπάρχει λόγος γι' αυτό. Φυσικά και ο Γερμανός Υπουργός έχει περισσότερο λέγει στα όσα αποφασίζονται. Επίσης ε, από αυτόν τον μήνακα προκύπτει ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν σχέση με το θέμα σας. πούμε τι γίνεται με την ε, διαφάνεια στην ε, νομοθεσία ή τέλο πάντων στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία και άλλα. Αν συγκρίνουμε επίσης το Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το κοινοβουλευτικό καλούπι βλέπουμε κάποια συμπληρωματικότητα. Όταν υπάρχει κοινοβουλευτικό στοιχείο σε κάποιο θεσμικό όργανο και αντιστρόφως διαπιστώνεται ότι υπάρχει αυτή η, το χαρακτηριστικό το ότι γίνονται συζητήσεις για να προχωρήσουν τα θέματα. Αυτό γίνεται στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Και όσον αφορά την διαφάνεια επίσης ε, δεν ισχύει. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την ε, κατανομή αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, αυτή την γελοφτική φύση του οργάνου. Βλέπουμε τώρα το τι θα πρέπει να γίνει παραπέρα για να κερδίσουν εμπιστοσύνη των ε, πολιτών, για να είναι πιο δημοκρατικά και σας τονίζω το ρίσκο, τον κίνδυνο του να έχουμε αυστηρή ε, υιοθέτηση των ε, χαρακτηριστικών του Κοινοβουλίου. Πλήρη, ας πούμε, διαφάνεια όσον αφορά τις ε, αποφάσεις. Επίσης, την ε, πολυσυλλεκτικότητα, τον πλουραλισμό στην εκπροσώπηση των κρατών μελών στα συμβούλια. Έτσι πάμε για γερουσία. Οπότε βλέπετε ότι αν έχουμε ε, μια μεικτή, ε, μια ήπια εφαρμογή των αρχών του Κοινοβουλίου. Έτσι μπορούμε να έχουμε συζήτηση σαν το Κοινοβούλιο σαν αρχή της διαδρομής κάποιου νομοθετήματος και στη συνέχεια όμως τα κράτη-μέλη να δηλώνουν την τοποθέτησή τους αυτά πριν τη λήψη αποφάσεως αλλά και αφού ληφθεί η απόφαση τότε θα είναι πιο αποτελεσματική η δημοσιοποίηση της απόφασης εάν γίνει ενημέρωση ε, κάποιο, με κάποιο δελτίο ε, προς εθνικά κοινοβούλια και μέσα ενημέρωσης. Παρακατώ τώρα βλέπουμε εδώ πέρα μια κριτική αξιολόγηση των ε, προτάσεών σας. Ας πούμε, πρώτα-πρώτα, για κάποια συγχώνευση των συμβουλίων, για την κυκλική εναλλαγή των προεδριών, όλα αυτά τα οποία τα πρότεινε πριν από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε σχέση με τα υπέρ και τα κατά είναι διαφορετικά βέβαια για Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Οπότε αυτό θα χαθεί αν αποκρίσει κοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά το Συμβούλιο. Επίσης, ένα άλλο βασικό θέμα είναι οι Υπουργοί. αν ασχολείται μόνο με την νομοθεσία, ε, τότε, το, το Συμβούλιο τότε δεν θα ε, πηγαίνουν στα Συμβούλια οι Υπουργοί και θα πηγαίνουν πρεσβευτές, ε, το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Επίσης, έτσι, θα καταλήξουμε στο να έχουμε Ε, παζάριμα γιατί θα ανταλλάσσετε το ναι σε μία πρόταση με το ναι σε μία άλλη. Τώρα όσον αφορά την διαφάνεια το Κοινοβούλιο θα συνεδριάζει ανοιχτά αλλά και το Συμβούλιο. Και σας προβλήμω στη συνθήκη του Μάστερ και τον κανονισμό του 2001. σε σχέση με τις διαδικασίες, τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν επομένω διάφορα νομικά στοιχεία και η αξιολόγηση βέβαια μοιραία είναι, καταλήγει σε μεικτά συμπεράσματα ότι για τη δημοσιότητα ε, θα είναι θετικό το αποτέλεσμα για τις ψηφοφορίες επίσης θα σταματήσει η ισχύουσα πρακτική ότι οι υπουργοί μπορούν να αποφύγουν να τοποθετηθούν και να υπάρχει λεγόμενη σιωπηρή πλειοψηφία. Εδώ θα έχουμε πρόοδο και αυτό αφορά και τα κάποια τέλο πάντων έγγραφα, κάποιε πληροφορίε για την Κορεπέρ. Και ε, αρνητικό θα είναι ότι στις πρώιμες φάσεις δεν θα υπάρχει διαφάνεια. Ε, δηλαδή στη φάση της Κορεπέρ και των ε, ομάδων του Συμβουλίου. Και για τους ε, τριμερείς διαλόγους θα έχουμε λιγότερες πληροφορίες. Επίσης θα θα γίνεται κατάχρηση του χαρακτηρισμού και της διαβάθμισης των εγγράφουν Επίσης, ε, έλλειψη κανόνων σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Και το ίδιο για τις τελικές ψηφορίες. Δεν θα υπάρχει ενημέρωση. Έχουμε την ε, του Transparency International και τη διαφάνεια έχουμε και άλλους ε, φορείς για τέτοιες αλλαγές για το ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, διαφάνεια να είναι πιο, πολλά έγγραφα διαθέσιμα και από την Κοζάκα έχουμε κάποιες τέτοιες προτάσεις ότι θα πρέπει ε, τρίμηνο η Κορεπέρ να παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Επίσης εδώ τονίζουμε τα εξής στην μελέτη μας. Θα πρέπει να προσεχτούν τα εξή, αυτά λέμε στην έκθεση. Πρώτα πρώτα ποιο θα είναι το τίμημα της ε, αποτελεσματικότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα λοιπόν και εάν υπάρχει περισσότερο φως στα όσα γίνονται στο Συμβούλιο τότε ε, υπάρχει ο φόβος ε, οι συνεννοήσεις, τα, τα, τα παζάρια συνεννοήσει να γίνονται αλλού, άτυπα, στους, διαδρόμου διαδρόμους ή αλλού. Και έτσι να υπάρχουν λιγότερες εγγύησεις ε, υπέρ των συμφέροντων των κρατών μελών. Κλασικό φιλοσοφικό θέμα ότι όταν ε, είναι πιο επίσημη, πιο τυπική μια οργάνωση, ένας οργανισμός, τότε επιδρά λιγότερο στο γίγνεσθε. Επίσης, λέμε παρακάτω για την ε, διαφάνεια όσον αφορά τις ε, κοινωνικές ιδιότητες. Ε, όμως, όταν συντριάζει για τους λόγους ένα κοινωνικό σώμα ε, και κλεισμένων, ε, τότε δεν έχει διαφάνεια. Έχουμε μάλλον εναλλαγή κάποιων φάσεων με πάρα πολύ διαφάνεια, όπως η Ολομέλεια, Έχουμε λιγότερη διαφάνεια σε άλλες φάσεις όπως σε συνδράσεις των επιτροπών και έχουμε επίσης και συνεδριάσεις που δεν έχουν καθόλου διαφάνεια όπως σε συνεδριάσεις κάποιων ομάδων βουλευτών, κάποιες συναντήσεις. Και νομίζω ότι είναι θέμα το κατά πόσο γίνεται σε κάποιο σώμα να υπάρχουν πλήρως αυτά τα χαρακτηριστικά του Κοινοβουλίου. Οπότε... Για το Συμβούλιο έχουμε την πρώτη φάση των συστάσεων και μετά έχουμε την, την επόμενη φάση που ψηφίζουν τα κράτη-μέλη Οπότε και γνωστοποιείτε το τι αποφάσισαν. Οπότε το μαθαίνετε και εσείς και το, και το Εθνικό Κοινόβουλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, Ραμόν. Να σας τα πω στα ισπανικά. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι συμφωνώ αρκετά με την κεντρική σας ε, ιδέα. Και δεν ξέρω μέχρι ποιου σημείου η Επιτροπή μας είναι υπέρ το Συμβούλιο να γίνει Κοινοβούλιο. Αλλά πάντως θεωρώ ότι τη σήμερα ημέρα με την κατάσταση αυτή της Ευρώπης δεν είναι ρεαλιστική μια τέτοια ιδέα. Δεν βοηθάει καν η Ευρώπη. Ίσως έχει ε, υπερβολική τάση λειτουργία λειτουργίας διακυβερνητικής. Κατά τη γνώμη μου, έχει ευξημένε υπερβολικές ε, εξουσίες Συμβούλιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυρίως. Οπότε όλα αυτά που όλα αυτά που αφορούν το επίπεδο το διακυβερνητικό, όλα αυτά να τα κάνουμε κοινοβούλιο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν στέκει και ούτε καν εξυπηρετεί. Και νομίζω ότι αυτό θα έφερε τις λειτουργίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα είχε πια η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν χώρο πολιτικού διαλόγου που τον χρειάζεται στο διακυβερνητικό αυτό επίπεδο. Οπότε Καλά, βέβαια δεν ξέρω ει βάθος, αλλά ε, τι, τι λέει αυτή η μελέτη, αλλά καταρχήν συμφωνώ. Και έχουμε τώρα το θέμα το άλλο, το θέμα της διαφάνειας. Αυτό είναι κάτι που το απαιτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Και αυτό επίσης όμως ε, θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο γιατί ακριβώ όπως λέγατε η διαφάνεια πολλές φορές η διαφάνεια έχει τίμημα λιγότερη ε, αποτελεσματικότητα. Ακόμα και όταν νομοθετούμε υπάρχουν κάποιες φάσεις στην διαδρομή της νομοθεσίας που αυτές οι φάσεις δεν έχουν διαφάνεια αλλά ε, που διευκολύνουν την διαδικασία, τη διαδρομή και έχω περάσει από ε, πολλά όργανα ε, κοινοβουλευτικά και έτσι γίνεται και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι μόνο είναι δυνατόν να αναζητούνται οι συνενέσεις. Εάν όλη η νομοθετική διαδρομή στο Συμβούλιο ε, χαρακτηριζόταν από διαφάνεια, τότε είναι σίγουρο ότι πάρα πολλές πολιτικές συμφωνίες που πρέπει να κλειστούν δεν θα ήταν ε, ε, εφικτές έχουμε, έχουν κάποιες τοποθετήσεις πολιτικές τα κράτη-μέλη ε, και μετά δεν μπορούν να κάνουν πίσω από αυτές με τη διαφάνεια. Τώρα για, να κλείσω. Ε, το θέμα είναι η σχέση μας με το Συμβούλιο. Ε, οι σχέσεις μας υλοποιούνται, ας το πούμε, στους τριμερείς διαλόγους. Εκεί ζητούμε τις ε, συνενέσεις και εκεί και έχουμε σημαντικές δυσκολίες. εδώ ε, είναι το θέμα που θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορούμε εδώ να εφαρμόσουμε τις ιδέες της πολιτικής επιστήμης για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους τρόπους για να διευκολύνονται, να έχουν αισιότερο τέλος ε, περισσότεροι τρίλογοι ε, για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, αυτό το μέτωπο είναι το πιο δύσκολο. Αυτά ήθελα να σας αναφέρω και φυσικά να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας κύριε Σίγητα. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσει από του συναδέλφου, θα ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι. Ιδίω σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί. Υπάρχει συνθήκη που προσδιορίζει και τις αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην πράξη έχει αλλάξει όμως τα τελευταία χρόνια η λειτουργία, ε, δεν πρόκειται μόνο για διαβούλευση και για ε, χορήγηση κατευθύνσεων για το μέλλον, αλλά πραγματικά παρεμβαίνει. Έχουμε την Προεδρία που έρχεται τον τριμερή διάλογο και λένε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν το κόμμα, γιατί είναι ε, ουσιαστικά εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην πράξη, λοιπόν, είναι διαφορετική κατεύθυνση. Όλο ένα και περισσότερες συμφωνίες δεν γίνονται από το Συμβούλιο των Υπουργών αλλά οι υπουργοί ε, μεταφέρουν το ζήτημα προς τα πάνω, προς ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε εντοπίσει αυτή την ανομοιογένεια μεταξύ ε, πρακτικής και συνθήκης. Ο Τζόρτζ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σας. Και εγώ θα ήθελα να θίξω το θέμα της διαφάνειας. Επειδή έχουμε υποστεί τεράστια πίεση ε, ως κοινοβούλιο για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Επομένω, εγώ να διερωτώ με ποιος είναι ο στόχο, στόχος τελικά. γιατί παρουσιάζεται η διαφάνεια ως εγγενώς καλή και ευκταία και ότι τα πάντα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο διαφανή. Αφενός, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ε, απεριόριστη ζήτηση για τη διαφάνεια. Αυτό θίγει ζητήματα δημοκρατικής αρχής εφόσον υπάρχει κάτι που είναι ε, άπειρο ή απεριόριστο, πώς μπορεί κάποιος να το ελέγξει δημοκρατικά. Είναι και φιλοσοφικό και πολιτικό ζήτημα. Δεύτερον, ε, η, η βάση, η αφετηρία αυτής της σκέψης είναι ότι υπάρχει καχυποψία απέναντι στην πολιτική. Οι δημόσιοι θεσμοί, κυβερνήσεις, και τεχνοκρατικές υπηρεσίες ε, δεν πρέπει να είναι... Ή μάλλον ε, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι 100% διαφανής, ενώ η μαλλον θεωρουμε οτι πρεπει να ειναι 100 διαφανης ενω και κοινωνια των πολιτών όχι, από την άλλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία στη δημόσια ζωή για το τι πρέπει να είναι διαφανές και τι όχι. Και αυτό θέτει και γύρει δύσκολα ζητήματα λογοδοσία. Παρακαλώ κύριε Ρόζενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ. για τα πρώτα σχόλια. Συμφωνούμε για αυτή την έλλειψη αποτελεσματικότητας με υπερβολική ενδεχομένως διαφάνεια. Ήθελα να επισημάνω το ζήτημα της ε, οικειοποίησης ε, των αποφάσεων από τους πολιτικούς. Αν έχουμε υπερβολικά πολλούς κανόνες, περιορισμούς, απόλυτες διαφάνειας, υπάρχει ο κίνδυνος οι πολιτικοί και οι ίδιοι οι υπουργοί να μην έρχονται καν στην ε, συζήτηση, να μην συμμετέχουν σε μια συζήτηση που έχει ε, ως στόχο την αύξηση και το περαιτέρω, την περαιτέρω εκδημοκράτηση της Ευρώπης. Μιλήσατε για τους τριμερείς διαλόγους. Θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω επισημοποίηση των τριμερών διαλόγων. Έχουν γίνει βέβαια προσπάθειες τα τελευταία δύο-τρία χρόνια να λάβουν μεγαλύτερη προβολή. Ξέρουμε ότι τα τρία θεσμικά όργανα προετοιμάζουν έναν ιστότοπο με μια βάση δεδομένων που θα δείχνει ε, την πρόοδο όλων των διαδικασιών. Εδώ και δύο χρόνια ξεκινήσει η διαδικασία, ελπίζω να ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι αυτή η επιγραμμική βάση δεδομένων θα βοηθήσει. Για τα σχόλιά σας, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ζήτημα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αποφασίζει αντί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Εξαιτία του κανόνα της ε, ομοφωνίας ή ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Και εναπόκειται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την κατάσταση και να επισημαίνει τα κακό κείμενα. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, όλο ένα και περισσότερο δίνει τον τόνο αντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μου φαίνεται πιο λογικό με βάση ε, τη μορφή που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κρίση. Τις, οι βασικές ε, αρχές λοιπόν και προτεραιότητες ε, δίνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό και κατανοητό, αλλά και πάλι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος. the EU level και βλέπουμε μια τάση από το 2010 και μετά μπορεί να συνδέεται με αυτό. Για το τελευταίο σας ε, σχόλιο, κύριε Σόφλιν, συμφωνώ με, τον, ε, με την αντίληψη ότι υπάρχει απεριόριστη ζήτηση ως προς το διαφάνεια και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος Τη διαφάνεια όμως δεν την πετυχαίνουμε μόνο με τους κανόνες και την ομολογία του δικαστηρίου, αλλά και μέσω ε, του ενεργού ρόλου των φορέων διαφανείας που ε, καταθέτουν ε, γραπτά ερωτήματα παράδειγμα μέσω του Κοινοβουλίου. Προκειμένου λοιπόν η επίτευξη της διαφάνειας δεν περνάει μόνο από τις κλασικές διόδους, αλλά και από τα μέλη των κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και λυπούμε για το γεγονός ότι δεν έχουμε παραπάνω χρόνο για να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα όταν προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε τις εκθέσεις μας, αλλά πραγματικά σας ευχαριστούμε γιατί τροφοδοτούν τα όσα ετοιμάζουμε και σε ό,τι αφορά το τομέα της διαφάνειας σε σχέση με την έκθεση του ε, διαμεσολαβητή. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό το σημείο τη ε, ε, ημερήσια διάταξη και περνάμε στο επόμενο και η κυρία Βος βρίσκεται είναι εδώ μαζί μας από την, το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ με την παρουσίαση που θα μα κάνει σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς της Ένωσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Oh yeah, there it is. Yeah. And the lady has disappeared, our colleague, dear oh, colleague, yes, who is doing it. No, but yes, it's, so maybe it's there. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο σας δεφάνες, πολύ ωραία. Καλώς. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακολουθήσω, να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της μελέτης που κάνουμε σε σχέση με τους οργανισμούς της Ένωσης. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχουν 36 οργανισμοί ε, τη σήμερα ημέρα ε, και εκκρεμεί και μία πρόταση για τη δημιουργία ενός ακόμα, δηλαδή της ε, Ευρωπαϊκής Οργανισμού Εργασίας και να πω ότι αυτό τα αυτοί οι οργανισμοί ε, είναι ε, πρόσωπα ενωσιακού δημοσίου δικαίου, αλλά είναι θεσμικά ξεχωριστά από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βρίσκονται δηλαδή κάπου ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δικό τους προπολογισμό και έχουν τη δική τους διοίκηση. Ο Μισελ και εγώ έχουμε αποκαλέσει αυτές τις, αυτούς τους οργανισμούς ως διαμεσολαβητές, in-betweeners, καθώς βρίσκονται ανάμεσα ακριβώς ε, στα θεσμικά όργανα αφενός και στα κράτη-μέλη αφετέρου. Ε, και θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα αργότερο. Οι οργανισμοί λοιπόν δημιουργούνται ως λύση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρίσεων και είναι ενδιαφέρον το, ε, το ότι παρατηρούμε αυτήν την, ε, τον πολλαπλασιασμό ε, των οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος αρχίζει να δημιουργεί ένα πρόβλημα ε, νομιμότητας από μόνο. Δηλαδή αρχίζει να, αυτός ο αριθμός των οργανισμών να αποτελεί πρόβλημα από μόνο του. Και ε, χαιρόμαστε για το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εστιάζει πλέον σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή των αποκεντρωμένων οργανισμών. Αυτό που κάναμε ε, ήταν καταρχήν να εξετάσουμε το πώ έχει η κατάσταση αυτών των αποκεντρωμένων οργανισμών σε σχέση με την κοινή προσέγγιση. Και εδώ εξετάζουμε για παράδειγμα τη βάση, τη λειτουργία του, τη χρηματοδότηση, τη σχέση με τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, του άλλου συναρμόδιου βαρύ και θα σας παρουσιάσω κάποια από τα πορίσματα αυτής της μελέτης ε, για να γίνει αυτή η συζήτηση. Ε, πρωτού περάσω στα πορίσματα, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει επισήμως αυτούς τους οργανισμούς κάνοντας συγκεκριμένες αναφορές ε, σε διάφορους οργανισμούς, ε, ό,τι αφορά για παράδειγμα την πρόσβαση ε, σε έγγραφα, τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ούτω καθεξής, αλλά εκείνο που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναφορά των οργανισμών σε άρθρα που θα αναμέναμε να αναφέρονται περισσότερο. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά τη κατεξουσιοδότηση και τι εκτελεστικέ πράξει, δηλαδή τα άρθρα 290 και 291 τη Ηθική τη Λισαβόνα. Ωστόσο, ε, στην ε, ε, περίπτωση της υπόθεσης ΕΣΜΑ ανοιχτή πώληση short selling το δικαστήριο ανέφερε ότι είναι διατεθειμένο να πληρώσει αυτό το νομοθετικό χάσμα των συνθήκων και μπορεί να και αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ε, οργανισμοί αυτοί μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν ε, στο πεδίο εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 τη συνθήκη. Άρα λοιπόν, όταν αναφερόμαστε σε αυτή την υπόθεση έσμα ανοιχτή πώληση, ε, τότε καλό είναι να θυμόμαστε ότι ουσιαστικά έγκυψε από την απόφαση του δικαστηρίου ένα νέο δόγμα μερώνει δύο, αν θέλετε. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες εξουσίες των οποίων χαίρουν αυτοί οι οργανισμοί αυτόνομες οι οποίες ε, μπορούν ε, να αφορούν για παράδειγμα σε πολιτικού, οικονομικού ε, και κοινωνικού χαρακτήρα αποφάσεις. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα πρέπει να εξετάσουμε την ανάληψη της ευθύνης από την πλευρά αυτών των οργανισμών της Ένωσης. Εξετάσαμε τώρα τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και των θεσμικών οργάνων αλλά και τη σχέση αυτών των οργανισμών με τα κράτη-μέλη και άλλους ε, αρμόδιους και σε ό,τι αφορά τη σχέση με ε, τα θεσμικά όργανα τη Ένωση και τα κράτη-μέλη, οι εν λόγω οργανισμοί ε, είναι πολύ ενεργοί στο πλαίσιο της θεσμικής δηλαδή δομής των θεσμικών οργάνων και αυτό καταδεικνύει βέβαια και τον υβριδικό του χαρακτήρα. Καθώς συμπεραίνουμε εγώ και ο Μισελ ακριβώς ότι λειτουργούν ως ε, ένα, ε, ε, ένα ενδιάμεσος εφορέας ανάμεσα δηλαδή στα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη και χρειαζόμαστε και περισσότερη έρευνα και μάλιστα θα υπάρξει μια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά την διοργάνωση μιας διάσκεψης ακριβώς σε σχέση με αυτό το ζήτημα, δηλαδή των σχέσεων αυτών των οργανισμών με τα κράτη-μέλη. Επίσης, το γεγονό τη θεσμική του ιδιαιτερότητα, δηλαδή ότι είναι χωριστεί αυτοί οι οργανισμοί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη, ε, σημαίνει ότι είναι ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα η ανεξαρτησία τους από επιρροή των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να απασχολήσει περισσότερο και εμά και γενικότερα την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι σχέσει των οργανισμών με του ε, συναμόδιου ε, φορεί, προβλέπεται ότι μπορούν να συμμετέχουν, για παράδειγμα, αυτοί οι οργανισμοί στα διοικητικά του συμβούλια και μπορούν να συνεργάζονται με τους οργανισμούς δηλαδή αυτοί οι φορείς ε, ε, στο πλαίσιο άλλων ομάδων, επιτροπών, δικτύων ε, με βάση τα όσα προβλέπει η κοινή προσέγγιση, το common approach. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολυμορφία συμμετοχής των συναρμόδιων φορέων όπως προβλέπεται στο ίδιο το καταστατικό των εκάστοτε οργανισμών. Εκείνο που επίσης αναφέραμε είναι ότι υπάρχει ε, ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά ε, τα εμπορικού χαρακτήρα συμφέροντα και βέβαια με τις ε, διαδικασίες έγκρισης του discharge, δηλαδή του προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε ακριβώς με τέτοιου είδους ζητήματα, δηλαδή σύγκρουση συμφερόντων και κάποια, κάποιοι κανόνες έχουν τεθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί και αυτό το ζήτημα. Και θα επανέλθω σε αυτό λίγο αργότερα. Τώρα, εξετάσαμε το ζήτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και είδαμε ότι υπάρχουν μία σειρά από διαφορετικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων το κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει έλεγχο σε αυτού του οργανισμού. Καταρχήν, μπορεί να το κάνει μέσω του διοικητικού του συμβουλίου, καθώ το κοινοβούλιο δικαιούται να διορίσει ένα μέλο αυτού του διοικητικού συμβουλίου και ε, είδαμε ότι πράγματι αυτό επιτρέπεται και από την κοινή προσέγγιση και διαπιστώνουμε ότι στις νομικές βάσεις των οργανισμών υπάρχει πολυμορφία και κατά συνέπεια σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχουν αμφιβολίε ω προ το κατά πόσο το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει ε, ένα μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον ασκεί έλεγχο και δημοσιονομικό ε, και επιχειρησιακό σε αυτού του οργανισμού. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή, δεν υπάρχει κάτι στην κοινή προσέγγιση, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι στι διάφορε νομικέ βάσει στα καταστατικά των οργανισμών υπάρχει ε, σωρία διαφορετικών ε, τρόπων ε, έγκριση των εκτελεστικών διευθυντών και στην πράξη ουσιαστικά η, η, ακριβώς υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση από αυτή που βλέπουμε στην κοινή προσέγγιση. Επίσης διαπιστώνουμε ότι τα πολυετή προγράμματα εργασίας επιτρέπουν την συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή και επίσης ε, υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις διαφορά απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ε, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις ε, απαιτείται μόνο η γνώμη από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ή σε άλλε περιπτώσει υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση μόνο του Κοινοβουλίου. Ενώ αντιθέτω η Επιτροπή προβλέπει σε αλλες περιπτωσεις υπαρχει υποχρεωση τη διαβούλευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, άπαξε ετήσιες ε, εκθέσεις. Υπάρχουν εδώ και σχετικές νομικές βάσεις σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και τη διαδικασία της ε, έγκρισης των προπολογισμών και ότι ε, πράγματι εξαρτώνται οι οργανισμοί αυτοί από τα κονδύλια της Ένωσης, οπότε πρόβλημα έγκρισης δεν υπάρχει, αλλά ε, το πρόβλημα προκύπτει για, τις αυτο, για τους αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς οι οποίοι δεν τίθεται σε κανένα είδους δημοσιονομικό έλεγχο του προπολογισμού τους δηλαδή. Επίσης υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικοί τρόποι ελέγχου και ε, ε, επαφές που υπάρχουν και αναφέρω εδώ ενδεικτικά για παράδειγμα ε, το ποια είναι αρμοδιότητα των εκάστοτε κοινοβουλευτικών επιτροπών σε σχέση με ποιου συγκεκριμένου οργανισμούς. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχουν επιτροπές οι οποίες έχουν αναλάβει δηλαδή στις αρμοδιότητες τους να εποπτεύουν περισσότερους οργανισμούς από ό,τι άλλες. Ε, επίσης εξετάσαμε τη, τη συνάφεια εδώ, δηλαδή το κατά πόσο έχει εφαρμογή στους οργανισμούς η κοινή προσέγγιση και διαπιστώσαμε ότι η συμμόρφωσή τους ε, δεν διαφοροποιείται πολύ κατά την περίοδο πριν το, την κοινή προσέγγιση ε, σε σύγκριση με την περίοδο μετά την κοινή προσέγγιση. Ε, διαπιστώνουμε δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όπως είπαμε σε ό,τι αφορά το διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στην νομική πρακτική των διαφόρων καταστατικών και νομικών βάσεων των οργανισμών. Ε, κάτι ακόμα που ήδη ανέφερα είναι το ότι συχνά δεν ζητείτε, ε, δεν απαιτείται διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό οφείλεται για παράδειγμα λόγω της κωδικοποίησης ή της φυστάμενης πρακτικής ε, ε, αλλά και λόγω της ετερογένειας της, των διαφορετικών οργανισμών και κατά την διαφορετική χρονική στιγμή της σύνταξη των σχετικών κανονισμών για την ίδρυσή τους. Κλείνω τώρα και έρχομαι στις συστάσεις ε, της ε, μελέτης σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα ε, την, την προσέγγιση, αλλά έχω και κάποιες συστάσεις γενικότερες σε ό,τι αφορά αλλαγέ των συνδικών, τις οποίες ωστόσο δεν θα αναφέρω εδώ. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η κοινή προσέγγιση διαθέτει κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και προσφέρει ένα ενιαίο, ενωπημένο όραμα σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς της Ένωσης, πράγμα το οποίο είναι αναγκαίο, αλλά χρειάζεται περισσότερη συνέχεια, ε, περισσότερη συνέπεια σε ό,τι αφορά τη δράση των ε, οργανισμών και ε, χρειάζονται περισσότεροι κοινοί κανόνες και διατάξεις. Αναγνωρίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα τον ετερογενή χαρακτήρα τους. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ωστόσο δεν θα ισχύουν για όλους τους οργανισμούς αλλά ενδεχομένω για συγκεκριμένες ομάδες οι κατηγορίες οργανισμών. Και αυτό ε, θα πρέπει να γίνει επανεξετάζοντας ταυτόχρονα τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα των διοργανικών ε, συμφωνιών όπως αυτές έχουν ε, συναυθεί και συζητηθεί στο παρελθόν. Μία ακόμα σύσταση θα ήταν να υπάρξει ένας ορισμός αυτών των οργανισμών γιατί όπως σας είπα εγώ εξέτασα 36 διαφορετικούς οργανισμούς ε, και ανέκυψε το ερώτημα του τι ακριβώς είναι ε, ο οργανισμός. Για παράδειγμα, ε, στα δίκτυα τα οποία τα οποία δημιουργούν οι ίδιοι οργανισμοί αναφέρονται για παράδειγμα σε 44 συνολικά συμμετέχοντες και καθώς συμπεριλαμβάνουν εκεί και τις συμπράξεις, τα joint undertakings οπότε θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό ορισμό προς το τι ακριβώς εννοούμε με τον οργανισμό. Επίση, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών, ε, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ρόλο και αν θα μπορεί δηλαδή να επιλέγει, να διορίζει ένα μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο ή αν θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιπρόσωπο από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω θα προβλέπετε στο καταστατικό, ή εάν θα πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα εμπειρογνώμονα όμως κάτι τέτοιο μπορεί να συνάδει με τον ρόλο τον ελεγκτικό που έχει απέναντι στον οργανισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ε, θεσπίσουμε ένα ε, ε, πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου από την πλευρά του Κοινοβουλίου και του οργανισμού και επίση θα πρέπει να ε, προβλέψουμε και κάτι σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων ε, πάντοτε στα πλαίσια τη συγκεκριμένη εντολή που έχει λάβει ο, ο κάθε οργανισμό. know, last one, sorry. Uh, I will... Okay, so this is the last one. Ωραία, τελευταία μου διαφάνεια λοιπόν. Τη Επίσης ε, θα πρότεινα ε, την αναδιάρθρωση των ε, μηχανισμών ανάπτυξη τη ευθύνης των οργανισμών γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπερφορτωμένοι οργανισμοί με υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτέ τι ευθύνε. και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο του να υπάρχει ακριβώς ε, αυτή, ε, ε, αυτή να είναι υπόλογοι οργανισμοί και στα κράτη-μέλη εφόσον για παράδειγμα δραστηριοποιούνται και διεθνώς εν οργανισμοί. Επίσης θα πρέπει να διατυπώσουμε συγκεκριμένους κανόνες σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμη διατάξεων που θα ισχύει για όλους τους οργανισμούς. Θα πρέπει να ισχύουν δηλαδή διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικές ομάδες. Ε, οργανισμών. Επίσης θα πρέπει οι ε, οργανισμοί αυτοχρηματοδοτούμενοι αυτή τη στιγμή να τεθούν υπό τον δημοσιονομικό έλεγχο, πράγμα το οποίο ήδη αντιμετωπίζεται εν μέρη ε, μέσω της κοινή προσέγγισης, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και πλέον θα μπορούσαμε να δούμε το κατά πόσο οι οργανισμοί οι οποίοι ακριβώς δρούν μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Νομοθεσίας εάν εφόσον έχουν ε, αποφέρουν κέρδη κατά πόσο ένα μέρος αυτών των κερδών θα πρέπει να επιστρέφει στον ε, ε προϋπολογισμό της Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος Γιώργης. Ευχαριστώ. Όλους ε, όσοι εργάστηκαν σε αυτό το θέμα και η παρουσίαση της κυρίας Βός με βοηθά ιδιαίτερα Προετοιμάσαμε αυτή τη μελέτη, εν μέρη βασιστήκαμε στο έργο της και εν μέρη βασιστήκαμε και, στην, ε, και στις διάφορες επισκέψεις που έκανα, όσο ήθιστε κιόλα. Αρχικά είναι θέμα δημόσιας δικυβέρνησης η άνθηση αυτών των ε, Ινστιτούτων και θεσμικών οργάνων. Η δυσκολία είναι πώς αυξάνεται η λογοδοσία όταν είναι ασαφής ο ορισμός ε, του οργανισμού αυτού καθ' αυτού. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυσκολία. Στην έκθεση λοιπόν ε, περιλαμβάνονται ορισμένε ε, συστάσεις για την εξομάλυνση αυτής της κατάστασης. Πρέπει να τα σκεφτούμε βέβαια Αυτά που είπε η κυρία είναι πολύ σωστά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της κοινή προσέγγισης. Προκειμένου οι οργανισμοί αυτοί να ακολουθούν μια σχετικά παρόμοια διακυβέρνηση πράγματι υπήρχε μια προσπάθεια διακυβερνητικής, διοργανικής μάλλον, συμφωνίας πριν από μερικά χρόνια, αλλά δεν προχώρησε. Η πρόταση που κατέθεσα εγώ στην προηγούμενη συζήτηση είναι ότι θα πρέπει να γίνεται ετήσια συζήτηση για τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών οργανισμών και πριν από αυτή τη συζήτηση να γίνεται και μία εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Πράγματι, οι οργανισμοί ε, υπόκεινται και μάλλον ε, ε, για τους οργανισμούς αυτούς ισχύουν οι ίδιοι κανόνες διαφάνειας και φυσικά για την τροποποίηση της συνθήκης. Εντάξει, εμείς μπορούμε να το ζητήσουμε, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να τεθεί στο ευρύτερο θεματολόγιο για την τροποποίηση της συνθήκης όπως ανέφερε η καθηγήτρια Βός, πρέπει να δούμε πώς ε, θα εγγράφονται αυτοί οι οργανισμοί ε, στη συνθήκη, κυρίως το 291 και 30 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από πλευρά μου. Έχω, έχω μείνει πέντε λεπτά για μια ζωηρότατη συζήτηση. The Commission was also willing to take the floor. Θέλει να πάρει το λόγο κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Να συγχαρούμε την κυρία Βός για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και τον εισηγητή κύριο Σόπφλινγκ για τις συζητήσεις που έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση αυτής της μερικής επιτυχίας που είχαμε μέχρι τώρα, ως προς την ε, υλοποίηση και την επίπεδο ε, των οργανισμών και των μοντέλων διακυβέρνησής τους με, τη με την κοινή προσέγγιση. Ωστόσο, παραμένουμε προσιλωμένοι σε αρχές όπως ε, η λογοδοσία, η αποτελεσματικότητα, Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πρόβλημα της ε, κοινή προσέγγισης. Μάλλον πρόκειται για έλλειψη βούλησης. Από πλευρά συνομοθέτη περισσότερο. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά βέβαια για το Συμβούλιο. Σε κάθε όμως ε, κλαδική νομοθεσία για τους οργανισμούς έχουμε επιμέρους ε, σενάρια και ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει λόγος που δεν είναι νομικά δεσμευτική η κοινή προσέγγιση, ακριβώς επειδή ήταν πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε σε αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι έχει κάποια προστιθεμένη αξία. Ε, οι διευθετήσεις ό,τι αφορά ε, τα κεντρικά του κάθε οργανισμού τις ευθύνες ε, των διοικητών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διεθνείς ε, δραστηριότητες των οργανισμών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς, αλλά υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Συμφωνώ πλήρως πάντως και με τους δύο μιλητές. Πρέπει να έχουμε, μάλλον κατά πόσο πρέπει να είναι πιο δεσμευτική ε, είναι μια πρόκληση αυτό. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία γιατί όταν καταρτιζόταν αυτή η πράξη ήδη ρύθμιζε πολλά διαφορετικά σενάρια και καταστάσεις. Αλλά πολύ συχνά γίνεται κατάχρηση ε, αυτής της ευελιξίας και τελικά τα πάντα επιτρέπονται όπως είπε η κυρία Βος. Δεν υπάρχει ε, λόγος να έχουμε 12 διαφορετικές διαδικασίες διορισμού ενός ε, διευθυντή, για παράδειγμα. Το Δεκέμβριο θεωρούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την έκθεση Σέφλινγκ και μετά πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Α, ξέρετε, δεν θα έχουμε διερμηνία σε λίγο. Μισό λεπτό να σας το πω και μετά. Ήθελα να σας πω, σε αυτή την κριτική σας αξιολόγηση, την κοινή προσέγγιση κλπ. Λάβατε υπόψη την προβολή του έργου των αποκεντρωμένων ε, υπηρεσιών ε, εκεί που βρίσκονται. Γιατί έχουμε όλους αυτούς τους καυγάδες για το πού θα πάει μια καινούργια υπηρεσία, πού θα μετακομίσει. Ποτέ, ποτέ όμως δεν έχουμε δει αυτού του είδους ε, του τι γίνεται επί τόπου, εκεί που βρίσκονται οι επικεντρωμένες υπηρεσίες. που αυτό που προβάλλουν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο, ως παρουσία. Αυτό ε, το λάβατε υπόψη στην ανάλυση σας. Να τα πούμε στα αγγλικά γιατί η διερμηνία θα σταματήσει. Σε ένα, δύο λεφτά στα αγγλικά. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπρέσο. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σέφλιν και την καθηγήτρια Φως για αυτή την ε, τόσο τόσο ενδιαφέρουσα μελέτη. Αυτά παράλληλα με τη δική μου και άλλων ε, προσπάθεια όσον αφορά την Επιτροπή. Οπότε είναι εκτελεστικέ πράξεις. Επίσης ένα άλλο θέμα που γίνονται από την Κομισιόν και αυτό γίνεται ε, εκτός του κοινοβουλευτικού ελέγχου όμως. Καλά, καλά, δεν έχουμε τώρα χρόνο να τα πούμε μετά με τον ε, κύριο Σέφλιν. Αλλά διαπιστώσαμε ότι γίνεται μια ομογενοποίηση όσον αφορά κάποιες από αυτές τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Και τα είπε η Επιτροπή για το προσωπικό και η λήψη αποφάσεων επιβάλλεται αυτό. Δεν θα έχουμε διερμηνία, οπότε... Α, θα, θα σας τα πω στα αγγλικά. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην πρότασή σας είναι Agreement. Δυστυχώς εδώ πρέπει να σταματήσουμε τη διερμηνία. But it could be done between the Parliament, the agencies and the Commission, for example, eventually the, the Council, also to ensure the problem of vertical